Θα αρχίσουμε λοιπόν σήμερα τη συνεδρίαση μα, Οι συνάδελφοι Κόξ και Βασνεύσκη έχουν καθυστερήσει. Γι' αυτό προτείνω να συνεχίσουμε κανονικά τη συνεδρίαση. Μετά έχουμε το διευρυμένο Προεδρείο και στις μία η ώρα ε, έχουμε τη συνάντησή μας, αλλά κάποιο αεροπλάνο έχει καθυστερήσει και οι δύο συνάδελφοι λείπουν. Ο συνάδελφος κ. Πουτικόφ θα πρέπει να κάνει χωρίς εμάς ε, το μεσημέρι. Και νομίζω ότι το προτιμάει, δεν θα κλάψει. Διαμαρτύρουμε, διαμαρτύρουμε. Το καθήκον υπερτερεί όλων. Λοιπόν, έχουμε τώρα τις ψηφοφορίες. Η, η πρώτη είναι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Δεδομένου ότι η κυρία Ρόμεν Όιτεν έχει επίσκεψη με έναν πρίγκιπα, θα το πάρουμε αυτό το θέμα ως πρώτο. Υπάρχει καμία παρατήρηση. Όχι. Οπότε θα ψηφίσουμε βεβαίως ηλεκτρονικά. Μία ψηφοφορία είναι μόνο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 34 ψήφοι υπέρ, 5 κατά ε, δεκτή. δεκτή η γνωμοδότηση. Και τώρα, όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, την ΑΕΒ, έχουν οι συγητές κάτι να προσθέσουν. Όχι, όχι. Ωραία. Ο Ρομπέρτο και εγώ Έχουμε συζητήσει επί μακρόν και με τους ε, συντάκτες των τροπολογιών, με τους ε, σκιώδεις κλπ. Και έτσι υπάρχει η Γενική Συμφωνία. Λοιπόν, ψηφίζουμε τροπολογία 1, συμβιβαστική, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε. Τροπολογία, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, τροπολογία 82 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ <clears throat> κατά αποχές ξανά παρακαλώ 87 υπέρ κατά Πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 87. Α, ναι, όχι, δεν ψηφίζουμε την εξαγωγή όπλων, ψηφίζουμε την ΑΕΔ. Όχι, δεν είναι το 10, είναι το 11, ΕΙΕΔ, Επιρρησία Εξωτερικής Δράσης. Ωραία. Ε, ε, πέραση της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά, αποχέ. δεκτή. 89 υπέρ. Κατά, αποχέ. απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 και 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 με την προφορική υπέρ κατά αποχές δεκτή 97-98 υπέρ κατά αποχές δεκτές Συμβιβαστική 5 με προφορική τροπολογία του κυρίου Κόβατσεφ. Υπέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Προτείνω μετά το security task να βάλουμε να καλύπτει γεγονότα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Covered events ε, outside of the EU. Έτσι ώστε να, έτσι κι αλλιώς είμαστε υπεύθυνοι. Να καλύψουμε λοιπόν και την έξω επικράτεια. Λοιπόν, συμβιβαστική 5 με αυτή την προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 100, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Α, απορρίπτεται διορθώνει ο πρόεδρο. απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά Κατά απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά Αποχέ απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά αποχέ, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά αποχέ. απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υποπρόεδρος καλύπτεται από την τροπολογία 1. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προχωρούμε στην 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κατο... Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. 124. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 125. Όχι, αυτή διευθετήθηκε. 121 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική 8. Ναι, εντάξει, Ρομπέρτο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεχνικό λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας. Από 1 έως 4. Ένα λεπτό. Στην 124 δεν, δεν αναλογεί με αυτό που ψηφίσαμε. 124. 1, 2, 4. Θα έπρεπε να είναι μείον. Α, τεχνικό λάθος λέει ο πρόεδρος. Εμείς είχαμε βάλει μείον, ενώ τώρα έχουμε εδώ το θετικό σήμα στην 124. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία. Επανερχόμεσα τώρα. 125 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 136 και 137 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτονται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 139, α, συμβιβαστική 10, συγγνώμη. Συμβιβαστική 10 με προφορική της κυρίας Γκόμες. Θέλουμε να προτείνουμε να προσθέσουμε αυτή τη μικρή αλλαγή παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των αντιπροσωπιών δέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα θέματα κλπ. κλπ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί τα δικαιώματα των γυναικών, λέει ο πρόεδρος, δεν καλύπτονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ νόμιζα ότι καλύπτονταν. Ε, ποιος λοιπόν συμφωνεί με την προφορική τροπολογία. Κατά, άποχες, δεκτή. Συμβιβαστική 10α. 10 bis. 10 α. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ε, τροπολογία 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 καλύφθηκε ε, 157-158 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται 129 υπέρ, είναι 59 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 161 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 130, 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 164 υπέρ κατά αποχές απο, απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 δις δύο φορές όχι 166 υπέρ 166 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 179 υπέρ δεν θεωρώ ότι ε, ε, η δικιά μου τροπολογία καλύπτεται από, το, την, 179, από την 178. Ο πρόεδρος, κοιτάξτε, αυτή η τροπολογία είχε συμφωνηθεί με, την, με τον... Ε, Und die Herr Kollege Saryusz-Wolski wir auch in der EVP-Fraktion haben. Με τον Kurt Balance. Και ε, το είχαμε κάνει αυτό σε συμφωνία με το ΕΛΚ. Αν θέλετε μπορούμε να ψηφίσουμε την 178 αν ο κύριος Σάρους Βόλσκι δεν καλύπτεται. Ωραία, λοιπόν, καλύπ... Ε, ψηφίζουμε 178. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. όχι λέει ο πρόεδρος, αποφασίσαμε, ψηφίσαμε. Πέραν του κανονισμού δεν υποχρονόμουν, αλλά ψηφίσαμε την τροπολογία σας και απερίφθη. Προχωρούμε. 179.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 των 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 191 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 191 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 23 ψήφοι υπέρ, 21 κατά, δεκτή, δεκτή. Κάποια κάρτα δεν λειτουργεί. Α, λέει ο πρόεδρος, έκλεισα τη ψηφοφορία νωρίς. Λοιπόν, πριν ψηφίσουν όλοι, ξανά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 191. Τρεις ε, λείπουν παρακαλώ, τρεις ψήφοι λείπουν. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, ωραία. 27 υπέρ, 21 κατά, δεκτή. Προχωρούμε. 192 τεχνικό ζήτημα, δεν ψηφίζεται. Κύριε Ντάφ, συμφωνείτε. 139 υπέρ, 193 συγγνώμη, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ε,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 20-21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, κατά, ένα λεπτό. 20, 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κα, 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33, 34, 35 συνέργεια εδώ, συνεργασία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50-51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 με την προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 59. Έληξε η ψηφοφορία. 19 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63-64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 dafür dagegen enthalten. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 7 να ελέγξω ηλεκτρονικά την 6. 6 παρακαλώ. Έληξε η ψηφοφορία. 23 προς 28 απορρίπτεται. 7. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. ΔΕΒΕ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 3. Υπέρ. Α, όχι 3. Δεβε 5. 5. ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ξανά ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ κατά 7 7 το 6 έχει καλυφθεί, η ΔΕΒΕ 6 καλύφθηκε. ΔΕΒΕ 7, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεκατρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται budget. Ένα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πέντε, budget, πέντε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντ, ένα,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 Πέρα της ψηφοφορίας, 38 ψήφοι υπέρ, 12 ψήφοι κατά, μία αποχή. Δεκτεί λοιπόν η πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα πάει στην Ολομέλεια? Μάλλον λόγω της έκθεσης της κυρίας Έστεν, η οποία μάλλον θα πάει το Μάιο, αυτή η έκθεση θα πάει τον Ιούνιο. Γιατί καλό είναι να τη συζητήσουμε η παρουσία της κυρίας Έστερν. Γι' αυτό θα έλεγα να πριν από τη συζήτηση, η παρουσία της ΥΠΑ της εκπροσώπου, να συναντηθούμε για να ολοκληρώσουμε, να, να βελτιώσουμε τυχόν μικροεκκρεμότητες, ε, μήπως τυχόν και δεν ψηφιστεί από τους φιλελεύθερους, να μπορέσουμε τέλος πάντων να χτίσουμε μία γέφυρα, ώστε να παρακολουθήσουμε σωστά την εξέλιξη του ζητήματος και να κάνουμε μία συνάντηση και μία κουβέντα πριν από την Ολομέλεια. Δεν Εγώ δεν συμφωνώ, ούτε βλέπω και το λόγο. Έχουμε συζητήσει προσεκτικά, έχουμε καταλήξει συμφωνία σε πολλά σημεία. Δεν αντιλαμβάνομαι διόλου την αναγκαιότητα της αναβολής και είμαι απολύτως και κάθετα αντίθετη. Πρόεδρος, κυρία Λέζινγκ, τον Μάιο δεν θα είναι παρούσα η κάθε άστον στην Ολομέλεια. Επειδή η έκθεση απευθύνεται στην ίδια, θέλουμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί της. Αυτό μου φαίνεται λοιπόν σκόπιμο ώστε να μην μένει κάπως μετέωρο. Και για τον λόγο αυτό έτσι θα, έτσι θα πράξουμε. Ορίστε εσείς κύριε Κοπά. On behalf of the we are again... Είμαστε κατά της αναβολής εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ορίστε. Στηρίζω την θέση της κυρίας Λόισινγκ. Δεν μιλούμε τώρα για την έκθεση της κυρίας Μιλούμε για την έκθεση Γκουαλτιέρη Μπροκ, εάν θα πρέπει να συζητηθεί τον Ιούνιο. Άλλο θέμα λοιπόν αυτό, τελείω. <laughs> τώρα θα έρθουμε στην αναβολή της έκθεσης Λέσινγκ. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην έκθεση για τις εξαγωγές όπλων. Ο κύριος Λίσεκ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πράγμα θέλω μόνο να πω για διαφόρους λόγους επειδή χρειάστηκε να έρθουμε πάλι σε επαφή με τις χώρες μέλη, γι' αυτό σκεφτήκαμε αν ίσως θα πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία. Όμως τώρα νομίζω εν τέλει ότι μάλλον τάσομαι υπέρ της ε, διεξαγωγής ψηφοφορίας τώρα. Ο πρόεδρος. Καλώς, ψηφίζουμε τότε. Κυρία Λόιζιν, έχετε... έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Προχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Η τροπολογία 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τσεκ λέει κάποιος. Τέλος. Απορρίπτεται με ισοψηφία 21-21. Τότε λοιπόν 66. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Α, 67. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά απορρίπτεται τώρα καλύπτονται οι υπόλοιπες 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Οι σοσιαλιστές ζητούν, ζητούν επαλήθευση. 73 λοιπόν, επαλήθευση. Τσεκ. Τέλος. 21 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται. 74-75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τέλος της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, επαλήθευση. Τσεκ. 84. Τέλος της ψήφου. 29 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε την επαλήθευση. Α, Α, όχι, Toolbox λέει ο Απερίφθη. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές αυτή χρειάζεται επαλήθευση ηλεκτρονικά. Πέρας. Εκτός και αν θέλει ο κύριος Πόσελτ. Επιμένει ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πόσελτ, μας τα χαλάσατε όλα. Εκατόν τέσσερα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι χαρακτήρα γλωσσικού περισσότερο 107-108 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 Τέλος 28 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση α όχι όχι είναι σαφής η απόρριψη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε επαλήθευση 22 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ Α, όχι, πρώτα 121. 121, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αυτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εδώ θα κάνουμε check συμβαστική 9 τέλος 22 υπέρ 24 κατά και 5 αποχές απορρίπτεται Α, όχι, μια στιγμή πρέπει να τις κάνουμε όλες τώρα. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έρχομαι τότε. 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131-32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται α 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά έλεγχος επαλήθευση Πέρας. Ψήφι 31 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με 22-24 α καλά καλά ας κάνουμε παρήθευση αλλά η πρόγνωσή μου είναι 22-24 και 5 αποχές πέρας 22 υπέρ 24 κατά και 5 αποχές. Είναι πάντοτε 29. Εξαρτάται αν θα πει ναι ή ECR. Ε, 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές τώρα το, αποτέλεσμα. 142 ξαναλέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149 υπέρ 149 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Οκ, okay, okay. υπάρχει προφορική τροπολογία, 154, προφορική τροπολογία 8 και μόλις ψηφίσατε ναι. Είναι για την παράγραφο 24α νέο. 153 έχει αποσυρθεί. Πρόκειται για λάθος το οποίο περιλαμβάνει η λίστα ψηφοφορίας που είχε διανεμηθεί νωρίτερα. 155 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 λέει ο πρόεδρος υπέρ Α156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση τέλος εγκρίνεται με ψήφους 27 υπέρ 20 κατά. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 αυτή εκπίπτει. Έρχονται τώρα ορισμένες ταυτόσημες. ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 170 έως 175 τροπολογίες Κρόνμπερκ. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί αυτές. Ωραία, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρα, τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 γλωσσικής φύσης. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εδώ επαλήθευση νομίζω ότι εγκρίνεται 25 Τέλος. Τελείως λάθος, τελείως λάθος τα είπα. Απορρίπτεται, όπως βλέπετε. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29-30 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική 3 υπέρ Α, χρειάζεται ε, να επανέλθουμε στην 43, την οποία δεν ψηφίσαμε. Ψήφι υπέρ τη 43. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Συμβαστική 3 λοιπόν. Πάλι. Εδώ με μπερδεύει διαρκώς ο γειτονάς μου. Κατά. Αποχές. Πάλι μου φαίνεται θα είναι το αποτέλεσμα 22-24. Πέρασε. Α, εγκρίνεται τούτη τη φορά. Με 24 ψήφους υπέρ, 23 κατά. Κάποιοι λιποτάκτες φωνάζει κάποιος. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 1 υπάρχουν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γλωσσικής φύσεως η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία ονομαστικά, ηλεκτρονικά δηλαδή Κυρίε και κύριοι, αν με είχατε ακούσει και είχαμε εγκρίνει την αναβολή, θα είχαμε γλιτώσει πολλή δουλειά. Και εσείς και εμείς. Απορρίπτεται λοιπόν η έκθεση και αρχιοθετείτε. Hmm? It's me, plus. <laughs> you know why? Because I have a plus If you want to know who was the... Αν θέλετε να γνωρίζετε ποιος ψήφισε υπέρ, ήταν ο κύριος Πάσκου. Διότι πάντοτε ακολουθεί την λίστα ψηφοφορίας της ομάδας του. Ήταν ο μοναδικός όμως. Αυτό θα πει πίστη στην κοινοβουλευτική ομάδα. The Australian Foreign Minister is coming any minute. Please stay. Καθίστε παρακαλώ, ο καλεσμένος μας έρχεται σε ένα λεπτό. Να είμαστε ευγενικοί, γιατί έρχεται από πολύ πολύ μακριά λοιπόν. In between I have to make a telephone call, you know, take over.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 Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση και καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας. Τον ευχαριστώ θερμά, τον καλωσορίζω που ήρθε εδώ μαζί μας και του δίνω αμέσως το λόγο.

Κύριε Μπροκ, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, είναι μεγάλη τιμή για μένα ω Υπουργό Εξωτερικών τη Αυστραλία να είμαι μαζί σα για να μιλήσω για την, ε, τις σχέσεις με την Ασία. Ή έχω την τιμή να έχω μιλήσει και στους πρέσβεις της Ένωσης στην Καμπέρα και τους είπα ότι η Αυστραλία και η Ένωση είναι φυσικοί εταίροι. Έχουμε κοινή δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου της ορθής διακυβέρνησης. Συντονίζουμε την απάντησή μας σε πολλές περιπτώσεις. Οι δύο πλευρές έχουν ε, άρει τους κυρώσεις μετά τις δημοκρατικές διαδικασίες του Μιανμάρ, για παράδειγμα. Συνεργαζόμαστε από κοινού για να ενθαρρύνουμε την ε, η νορθή διακυβέρνηση, καλή κυβέρνηση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την, ενώ ταυτόχρονα η περιβαλλοντική επίγνωση είναι αποτέλεσμα κοινή μελέτης από πλευράς μας. Είμαστε λοιπόν φυσικοί εταίροι και γι' αυτό είναι εντυπωσιακό το ότι η Αυστραλία με έναν ευρωπαϊκή καταγωγή πληθυσμό δεσμεύθηκε πέρυσι να αποκτήσει άνευ προηγουμένου σχέσεις με την Ασία. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Αυστραλία θα κερδίσει λόγω και της γεωγραφικής της θέσης από μια βαθύτερη εμπλοκή στην συνεργασία με την Ασία σε αυτό τον ασιατικό αιώνα. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ σε εσά είναι ότι η επανάσταση που γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια στην Ασία δεν είναι μόνο οικονομική μεταμόρφωση. Ω οικονομική μεταμόρφωση αποτελεί μία από, την ταχύ, μία από τις ταχύτερες μορφές εξυγχρονισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα ωστόσο συνιστά και μία κοινωνική επανάσταση, θετική συνολικά. Πριν από 30 χρόνια στην Ινδονησία, μόνο τα δύο τρίτα των παιδιών ολοκλήρωναν τη δημοτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, σήμερα κάθε παιδί σχεδόν βγαίνει από το δημοτικό. Το 2009 ένας στου 20 ιστορικά διορθώνει ο μιλητής, ένας στους 20 φοιτητές στην Ταϊλάνδη, την, τις Φιλιππίνες έβγαινε από το Πανεπιστήμιο. Τώρα το, ο συντελεστής αυτός είναι ένας στους τέσσερις. Όλο και περισσότερα πανεπιστήμια της Ασίας μπαίνουν στα ανώτατα πανεπιστήμια του κόσμου. Το 2000 η πολιομιελίτιδα εξεριζώθηκε από το Βιετνάμ. η μείωση της παιδινικής θνησιμότητας είναι από το 63 στο 23. Η στην ισότητα των ε, φίλων, το 1999 στην Καμπότζη μόνο 53 κορίτσια πήγαιναν στο γυμνάσιο για 100 αγόρια. Στην Καμπότζη, μία από τις πιο φτωχές χώρες στην Ασία ακόμα και σήμερα, η σχέση είναι 82 με 100. Στην Κίνα το 1991 75 κορίτσια πήγαιναν στο γυμνάσιο για 100 αγόρια. Τώρα είναι περισσότερα τα κορίτσια στο σχολείο από τα αγόρια. Στην, ε, στις Φιλιππίνες, στην Ταϊλάνδη, στην Κίνα υπάρχουν πλέον περισσότερες φοιτήτριες από ότι φοιτητέ. Η Ασία αλλάζει τα τελευταία 50 χρόνια. Μεταμορφώθηκε και δεν αφορά αυτό την Κίνα μόνο και το τονίζω στην Επιτροπή σας. Πολλές άλλες αφηγήσεις υπάρχουν. Η Μογγολία, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο. Η ανάπτυξη προβλέπεται φέτος να, να ξεπεράσει το 15%. Μια χώρα που αποφάσισε στη δεκαετία του 90 ε, ε, συνειδητά να γίνει πολυκομματική δημοκρατία, να επιτρέψει δηλαδή στον κόσμο, να στους πολίτες να αποφασίσει την επιλογή της κυβέρνησης. Οι αλλαγές κυβερνήσεων μαρτυρούν αυτό και το αναγνωρίζει αυτό συμβαίνει όπως θα συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα από εσά. Να η Μογγολία, άλλη αφήγηση, η Ινδονησία, μία mainstream μουσουλμανική χώρα εμπιστεύεται τους πολίτες να επιλέξουν την κυβέρνησή τους με πολυκομματική δημοκρατία, ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, πρόεδρο ε, υπόλογο σε ένα ισχυρό κοινοβούλιο με δημόσιο διάλογο για τα θέματα διακυβέρνησης, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, με στρατιωτικές και αστυνομικέ δυνάμεις υπόλογες τους πολιτικούς, χώρα που παροτρύνει και πιέζει άλλους να παρακολουθήσουν, την, να περιορίσουν το ρόλο του ε, στρατού, τονίζοντας ότι η θέση του στρατού είναι στα στρατόπεδα. Η Ινδονησία έχει ακολουθήσει πολιτικές αντίστοιχες με τις Ευρώπης. Ε, η ειρηνική επίλυση συνοριακών διαφορών, επιστροφή του στρατού στο στρατόπεδα. Ενώ είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα. Τέτοιες αφηγήσει βρίσκουμε πολλές. Η Ιαπωνία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δύναμη της δημοκρατίας στην Ιαπωνία το ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ε, σήμερα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της χώρας. Η Ιαπωνία είναι συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες μείωσης των ανθρωπιστικών καταστροφών στον κόσμο. Είναι μια ζωτική, συνεχιζόμενη δημοκρατία. Είδε σειρά αλλαγών κυβερνήσεων χωρίς πρόβλημα. Για μας την Αυστραλία είναι η σημαντικός εταίρος και επαναλαμβάνω τονίζω ότι υπάρχουν πολλές αφηγήσει αυτής της επανάστασης που βιώνουμε στην Ασία. Ως Αυστραλία αναγνωρίσαμε ότι η Ασία παράγει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής. Σύντομα θα καταναλώνει 50% της ε, παραγωγής. Αυτό δείχνει την ανάπτυξη, την αύξηση και την γένεση στην Ασία μιας μεσαίας τάξης. Ένα κομμάτι της επανάστασης της Ασίας. Το 2030 θα υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια μέσω μέσοαστοί καταναλωτές στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού. Και υπάρχει μια δημογραφική δυναμική εκεί. Στην Ινδονησία, στην Ινδία το 2020 η μέση ηλικία τη Ινδία θα είναι 29, ένα, μια δυναμική δημογραφική ασύλληπτη. Αυτό είναι μια θετική πορεία. Να σας δώσω ωστόσο και μια αξιολόγηση που λέει ότι η πορεία αυτή έχει δύο, ενέχει δύο κινδύνους. Χώρες που ακολουθούν την πορεία της Ταϊβάν, της Κορέας, της Σιγκαπούρης, της Ιαπωνίας νωρίτερα, εκβιο, εκβιομηχάνηση, εκδημοκρατισμός, αλλά υπάρχουν δύο κίνδυνοι σε αυτή την πορεία. Πρώτον, η παγίδα του μεσαίου εισοδήματο, Δηλαδή, ότι τα προβλήματα της διακυβέρνησης, Φερρυπίν, διαφθορά, τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, θα εμποδίσουν τις χώρες να περάσουν από μέσου εισοδήματος χώρες σε υψηλού εισοδήματος χώρες χωρίς δηλαδή να υπάρξουν ε, σημαντικές ε, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Δεύτερος κίνδυνος, και αν θέλετε να σας παραπέμψω και στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Κίνα 2030, που λέει ότι η οικονομική απόδοση της Κίνας ήταν μια μοναδική success story, επενεί την Κίνα για την ενσωμάτωση της στον κόσμο, την προσαρμογή της στις νέες τεχνολογίες, την υποδόμη, τη δημιουργία παγκοσμίου επίπεδου υποδομών, αλλά ταυτόχρονα η, έκθεση την οποία εν μέρη πλήρωσε και η Κίνα ζητά να υπάρξει μια άλλη σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Κίνα για να ενισχυθούν τα θεμέλια μιας οικονομίας της αγοράς μέσω της ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων και της εφαρμογής συστημάτων νομικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Προειδοποιεί ότι, ότι αυτό πρέπει να το κάνει Κίνα για να, η Κίνα για να αποφύγει το να μείνει στην, στο χώρο των, μεσαίων, των χωρών μεσαίων εισοδημάτων. Αυτό το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες της περιοχής. Προκλητικές μεταρρυθμίσεις και κίνδυνος να μην προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις λόγω των κεκτημένων συμφερόντων. Άλλη πρόκληση, η δεύτερη πρόκληση σε αυτή την θετική αφήγηση ανάπτυξη σε όλη την Ασία είναι η πρόκληση που, θέτει, που θέτουν οι κίνδυνοι ασφάλειας λόγω εδαφικών διαφορών. Είδαμε τις διαφορές αυτές στην θάλασσα της Νότιας Κίνας και στην θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Η Αυστραλία δεν παίρνει θέση σε αυτές τις εδαφικές διαφορές, αλλά ζητούμε να υπάρξει ρύθμιση βάσει του διεθνούς δικαίου και μεταξύ άλλων της ε, Παγκόσμιας Σύμβασης του ΟΗΕ για, την, για το δίκαιο της θαλάσσης. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πάρα πολλά αν πετύχουμε συμφωνίες κοινή εκμετάλλευσης θαλάσσιων πόρων μεταξύ των χωρών ε, που, των, των, των χωρών που βρίσκονται σε σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η επίλυση της διαφοράς για θέματα κυριαρχίας νησιών και η σύναψη συμφωνιών για την ανάπτυξη και καταμερισμό της εκμετάλλευσης και των κερδών των πόρων είναι θετικό. Τρία προηγούμενα υπάρχουν στην περιοχή της Νότιας Κίνας για συμφωνίες ε, καταμερισμού των πόρων. Πρώτον, διαφορές μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ, μεταξύ Κίνας και Φιλιππινών και Κίνας και Μπρουνέη. Αυτές οι συγκρούσεις, οι διαφορές είναι ανησυχητικέ. Ε, μπορεί να δημιουργήσουν παρανοήσεις και τη χρήση βίας. Το ίδιο ισχύει και για, τις, ε, τη διαφορά μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας για το, τα νησιά Νταέγου Σενκάκο ή Σενκάκο. Ζητούμε να υπάρξει διάλογος στη θάλασσα της Νότιας Κίνας για να εξεταστεί η βιωσιμότητα συμφωνιών καταμερισμού των πόρων αντί να τρογόμαστε με θέματα κυριαρχίας. Εμείς η Αυστραλία είμαστε σύμμαχος με τη ΣΥΠΑ, αλλά η σχέση μας με την Κίνα αυξάνει σε σημασία. Πριν από δύο εβδομάδες η Πρωθυπουργός της Αυστραλίας συνήψε με τον Πρωθυπουργό κύριο και τον Πρόεδρο Τζι συμφωνία για μια στρατηγική εταιρική σχέση. Μεταξύ των οποίων είναι μια εγγύηση συνεδριάσεων σε επίπεδο κορυφής σε αιτήσια βάση. Επίσης, να τονίσω κάτι που είπε ο Πρωθυπουργό τη Σιγκαπούρη, ο Λί Γιού, ο οποίο είπε ότι η ασφάλεια στην ε, Νότια Ασία μπορεί να αποκτήσει ένα ξενοφοβικό χαρακτήρα αν δεν γίνει κοσμοπολιτική, διεθνής και εξωστρεφής. Οι δύο αυτές εναλλακτικές της ανάπτυξης της Κίνας είναι εξίσου πιθανές. Δεν υπάρχει τίποτα το αναπόφευκτο να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύουμε ως σύμμαχοι των ΗΠΑ, ως ισχυροί εταίροι της Κίνας, ότι η άνοδος της Κίνας είναι καλή για την Κίνα και καλή για τον κόσμο. Και, ο, και η λέξη ανάσχεση δεν έχει θέση στη, στο διπλωματικό λεξιλόγιο τον ΙΠΑ της Αυστραλίας ή άλλων. Η εμπλοκή με την Κίνα και της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι θετική και για μας και για τον κόσμο. Μια ισχυρή αμερικανική παρουσία στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού και μια ισχυρή συμμαχία μας είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε την συνέχιση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή. Τώρα, για τη Βορειοανατολική Ασία και τα προβλήματα στην Κορεατική ε, Χερσόνησο. Η αμερικανική παρουσία τα τελευταία χρόνια εκεί ήταν το θεμέλιο της ειρήνης και της Αφαιρότητα, Η παρουσία των ΗΠΑ σήμερα είναι σημαντική για να παράσχει εγγύηση προς την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα που αντιμετωπίζουν την πολεμοχαρή στάση της Βορείου Κορέας. Κλείνω μιλώντας για το ΑΣΕΑΝ και την μεγάλη σημασία του. 500 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμό των 10 χωρών του ΑΣΕΑΝ. Υπογραμμίζουμε τον κεντρικό ρόλο που παίζει στην ε, περιοχή και που αναγνωρίζουμε εμείς. Θα ενισχύσουμε την δραστηριότητα εξωτερικών σχέσεων. Η... Το ΑΣΕΑΝ είχε δίκιο για το Μιανμάρ πριν η Ευρώπη αναγνωρίσει την, το βάθος των αλλαγών. Το ΑΣΕΑΝ, το ο Οργανισμός Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ασίας, έλεγε ότι οι μεταρρυθμίσεις του πρόεδρου Τεντσέιν θα ήταν χωρίς επιστροφή. Ότι γινόταν κάτι σημαντικό στη χώρα αυτή. Ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει κινδύνους για να ξαναγυρίσει το στρατό στα στρατόπεδα και για να ακολουθήσει την πορεία του εκδημοκρατισμού. Πέρυσι το καλοκαίρι είχα πάει στο Μιανμάρ και είπα στον πρόεδρο Τιντσέιν ότι η Αυστραλία ήρε, δεν ανέστελε απλά τα, τις κυρώσεις. Και από ό,τι είδα χτες η Ένωση αποφάσισε να άρει τις ε, κυρώσεις κατά της χώρας. Είχαν δίκιο λοιπόν το ΑΣΕΑΝ στον, Μιανά, Μιανμάρ γιατί βρίσκεται στο κέντρο της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ενοποίησης της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η περιφερειακή συνεργασία είναι κλειδί για να εξασφαλίσει ότι αυτή η πορεία ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική Ασία, σε όλη την Ασία θα έλεγα, θα συνεχιστεί προς όφελο, όλων, μειώνοντας τις ανισότητες, τις ανισότητες μεταξύ φύλων και, το προσδόκιμο, και αυξάνοντας το προσδόκιμο ζωής. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου δώσετε να απευθυνθώ σε εσά και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις που θα θέσετε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών για την ε, θαυμάσια εισαγωγική σας ομιλία. Και η ευκαιρία αυτή είναι εξαιρετική διότι μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε αυτήν ε, την ήπειρο ή αυτή την πλευρά του κόσμου από μία άλλη οπτική γωνία. Ας συνδυάσουμε τώρα τη συζήτηση αυτή και με τη συμφωνία πλαίσιο η οποία τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, σε καλή εξέλιξη θα έλεγα, αλλά θα έλεγα ήθελα να ζητήσω την άδειά σας για να διακόψουμε λίγο μου, μου είπαν ότι η, η κοινότητα των μαρονιτών στον, ε, στη Συρία θέλει την υποστήριξή μας διότι απήχθη ο επίσκοπος με τον Ορθόδοξο επίσκοπο εκτελέστηκε ο οδηγός και ο σωματοφύλακας και εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα εξ ονόματό σα να έρθω σε επαφή με την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης και να εκφράσω την αγανάκτησή μας για αυτήν την κατά την απαγωγή, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά. Η κυρία Γκόμες ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Υπουργέ, με μεγάλη χαρά άκουσα τις απόψεις σας και συμμερίζουμε και εγώ την, ε, ε, τις αναλύσεις σας για τα θετικά ε, στοιχεία αλλά και για τις απειλές ε, στην περιοχή αυτή του κόσμου. Έχω και εγώ τις απόψεις μου και θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, ξεκινώ από την ανάλυση τη δική σας. Θα λέγατε ότι η Κίνα μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μία φούσκα, να υπάρχει μία φούσκα σε εξέλιξη η οποία σύντομα θα σκάσει και η οποία θα απειλήσει βεβαίως ολόκληρη την περιοχή, όχι μόνο την Κίνα και τους πολίτες της. Πώς ε, επίσης κρίνεται την αντίδραση, την, η, την έλλειψη αντίδρασης ε, της Κίνας ε, στα γεγονότα της Βορείου Κορέας, δεδομένου ότι είναι σύμμαχοι και πώς πιστεύετε ότι, τι θα γίνει με την περιοχή αυτή με, λόγω της συμπεριφοράς αυτής της Βορείου Και επίσης θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Ε, αναφέρετε τη Σιγκαπούρη, ε, το Χονγκ Κόνγκ, είπατε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι πιο σημαντικοί φορολογικοί παράδεισοι στον κόσμο και ιδιαίτερα για τους ε, ε, ενδιαφερόμενους για τους, ε, της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα, πιστεύω λοιπόν ότι και εσείς ανησυχείτε για αυτή την εξέλιξη η οποία σημειώνεται και είναι υπεράνω του νόμου. Είναι βεβαίως παράνομες αυτές οι ενέργειες αλλά είναι υπεράνω του νόμου όλες αυτές οι ενέργειες για τους φορολογικούς παραδείσους. Αναφέρεται λοιπόν αυτή την διαδικασία για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία. Είδαμε θαυμάσιες εξελίξεις στην Ινδονησία. Ε, δεν βλέπουμε δυστυχώς όμως τις ίδιες εξελίξεις στην Κίνα. Το Μιανμάρ, πρώην Βιρμανία, αναφέρατε τις αλλαγές που έχουν γίνει και τις οποίες προέβλεψε κατά κάποιο τρόπο η οργάνωση του ΑΣΕΑΝ. Είναι η κυβέρνηση έτοιμη να απορρίψει την Κίνα, αλλά μήπως υπάρχει ο κίνδυνος λόγω ορισμένων αλλαγών, παραδείγματο χάρη είσοδος της Σαν Σαν στο Κοινοβούλιο, διακυβεύει τη δημοκρατία ή την ενισχύει. Πώς κρίνεται την ε, στάση της Αγ ε, Τσι σε σχέση με τις μουσουλμανικές ε, μειονότητες, τους Ρουίντας και την καταπίεσή τους. Και πώς το Ανατολικό Τιμόρ, επίσης, μεγάλη επιτυχία. Εσείς παίξετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε εξελίξη εκεί. Πώς έχουν εξελιχθεί οι διαβουλεύσεις σας με το Ανατολικό Τιμόρ. Έχετε τίποτα καινούργια να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Να είσαστε λίγο πιο σύντομοι από την Άννα, η οποία ξέρει πάρα πολλά, ε, αλλά αν μπορείτε να συντομεύετε. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λέει ο μιλήτρια. Πρόεδρε, εσείς είστε πάντοτε λακωνικός και θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το παράδειγμα σας. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας και για την ανάλυση σας. Δεν θα σας ε, παρουσιάσω την ιστορία της ζωής μου, αλλά ο σύζυγός μου και εγώ έχουμε κυβερνήσει, έχουμε, συγγνώμη, ταξιδέψει εκτενώς στην Νοτιοανατολική Ασία. Έχουμε επισκεφθεί πολλές χώρες, πραγματικά εκτενώς πάντοτε προσπαθούσαμε να διαβάζουμε τις τοπικές εφημερίδες στα αγγλικά, διότι βεβαίως στις άλλες τοπικές στις ε, τοπικές διαλέκτους και γλώσσες καταλαβαίναμε. Διαβάζαμε λοιπόν τα αγγλικά νέα και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάσαμε, ε, οι καλές κριτικές, οι καλές κρίσεις, οι θετικές κρίσεις για τον Chris να αποτελούν προσβολή για τους Κινέζους λόγω της ε, κυβέρνηση της θέσεως στο Χονγκ Κόνγκ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, πώς ε, εξελίχθηκαν οι προσπάθειες της δικιάς σας κυβέρνησης για τη βελτίωση των σχέσεων με, τις, ε, με τους σημαντικούς εταίρους της, των νοτιοανατολικών ασιατικών χωρών. Καταλαβαίνω ότι καταβάλλετε μεγάλες προσπάθειες. Ορισμένες χώρες έχουν δημοκρατικά καθεστώτα, αλλά ορισμένες έχουν πολύ αρνητικά άσχημα δικτατορικά ιστορικά καθεστώτα. Παραδείγματος χάρη Καμπότζη, η οποία καταδιώκει και καταπιέζει ε, τους, ε, την αντιπολίτευση σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη, η άποψη της κυβέρνησής σας όσον αφορά την Ταϊουάν υποθέτω ότι υποστηρίζεται την πολιτική μια ενιαία Κίνα. αλλά στην πρακτική εφαρμογή τώρα, ρεαλιστικά, πώς αξιολογείται τη σημασία της Ταϊουάν εν σχέση με τις εξελίξεις στην θάλασσα της Νότιας Κίνας. Θα με ενδιαφέρει πολύ η άποψη την άποψή σα. Είχα τη χαρά να επισκεφθώ και τη δική σας χώρα όταν κάνουμε όλα αυτά τα ταξίδια με τον άντρα μου. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και μένω με χαρά τι απαντήσει σα. Ο πρόεδρο. Η κυρία, Θεοχάρου. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας. Επιτρέψτε μου να πω πόσο θαυμάζω το έθνο της Αυστραλίας και τον ε, ρόλο της ε, στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού από την οποία έχω προσωπική εμπειρία λόγω της ζωής μου εκεί. Η Αυστραλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην, ε, διαμόρφωση και στην ενίσχυση της και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής και στην Κύπρο ακόμα ο, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών είναι πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας. Δεν θέλω να θέσω ερώτηση, θέλω να εκφράσω την επιθυμία μου για μια επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και υπόσχομαι ως εισηγήτρια να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω στην ολοκλήρωση του στόχου αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιουτικόπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η πρώτη μου ερώτηση αφορά την ανάλυση σας για τον αντίκτυπο του κομβικού λεγόμενου ρόλου τον είπα στην, ε, στον Ειρηνικό και στο ΑΣΕΑΝ. Εγώ πιστεύω ότι με τις πρόσφατες ε, κινέζικες κινήσεις φαίνεται ότι ολόνα και περισσότερο υπάρχει μία σύμπτωση κινήσεων ε, που πιέζουν την συνοχή του ΑΣΕΑΝ. Δεύτερη ερώτηση. αφορά τις, Αυστραλο... τις σύνοαυστραλικές σχέσεις. Λέτε ότι είναι στρατηγική σημασία. Στηρίζεται σε αξίες, σε συμφέροντα. Ποια είναι η βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Αναφερθήκατε στον Κουαν Γιο, ο οποίος ε, στην παράθεση που αναφέρεται δείχνει ή μάλλον φαίνεται να δείχνει ότι η εξέλιξη του κινέζικου ρόλου εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο η Δύση σχετίζεται με την Κίνα. Συμφωνείτε με την ανάλυση αυτή. Δεν υπάρχει κινέζικη προέλευση της κινέζικης συμπεριφορά, δηλαδή αντικατοπτρίζει απλά την στάση των άλλων. Είπατε ότι είναι καλή η άνοδος της Κίνας για πόσο καιρό θα παραμείνει και πόσο καλή αν η εξωτερική πολιτική της Κίνας ε, αποκτήσει όλο ένα και πιο αυταρχικό κατηγορηματικό χαρακτήρα. Επίσης, μπορείτε να σχολιάσετε τις αλλαγές της εξωτερικής συμπεριφοράς ε, της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας για φερειπίν ε, το πρόβλημα των νησιών Σενκάκο ή Νταεγού. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σπάνια έχουμε εκπροσώπους της κοινοπολιτείας στην Επιτροπή μας. Τρεις είναι οι χώρες της κοινοπολιτείας της Ένωσης, αν ε, δεν το κατασκεφτεί. Πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου, η Κύπρος και η Μάλτα. Όπως ξέρετε, η Νότιος ε, Κορέα και η Σιγκαπούρη ήδη έχουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Ένωση, ενώ συζητείτε μια τέτοια συμφωνία με την Ιαπωνία. Θα κάνετε κι εσείς μια τέτοια συμφωνία ως Αυστραλία. Επίσης, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ιδίω ε, στον τομέα της καταπολέμησης της πειρατεία στα ανοιχτά της Σομαλίας. Υπάρχει η επιχείρηση Αταλάντη της Ένωσης. Θέλει να εμπλακεί σε αυτήν η Αυστραλία τι ρόλο θέλει να παίξει. Θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Καλή είναι και προφανώς η Αυστραλία θέλει να καταπολεμήσει τη διεθνή τρομοκρατία γιατί ήταν και θύμα ε, στην, στο, στις βόμβες στον Παλίο, στην Ινδονησία. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε ήδη στους Ροχίνγκια. Ε, εξωτερική πολιτική τώρα. Μιλήσατε για το θέμα της, του μοιράσματο των πόρων. Ε, ε Έχετε δει το σχέδιο του Προέδρου Μάε, της Προέδρου Μάε στο Ινταϊβάν ε, που μιλάει για να, ξεχωρίσουμε τις διεκδικήσεις ε, ιδιοκυριότητας και τις διεκδικήσεις ε, εκμετάλλευση κάτι όπως αυτό που έχουμε στην Ανταρκτική. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε στην περίπτωση των Σενκάκου να υπάρξει μια αντίστοιχη εκμετάλλευση. Κάτι άλλο, πώς είναι οι σχέσεις σα με την Ινδία. Άλλη μεγάλη χώρα της κοινοπολιτεία στην Νότια Ασία. Είναι ισχυρε πόσο ισχυρε είναι. Τελευταίο θέμα. Ανατολικό Τιμόρ. Είδα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ που κατηγορεί την Αυστραλία, αυστραλιανές εταιρείε μάλλον, για εξόριξη offshore ε, πετρελαίου χωρίς να πληρώνουν ε, την απαραίτητη, τα απαραίτητα royalties. Ε, πώς πάει η συνεργασία μεταξύ Timor Leste και Καμπέρα για το θέμα της καταβολής του τιμήματος από τις εταιρείε που κάνουν εξόριξη offshore. Ο κύριος Φως, αντιπρόεδρος τη Αντιπροσωπείας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας του ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας, τις αναλύσεις σας. Σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου μόνο στην, στις εξωτερικές σχέσεις, αλλά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας. Ε, κάνουμε τακτικές συνεδριάσεις, τακτικές συναντήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Αυστρα... Ε, ε, Κοινοβουλίου της Αυστραλίας από το 1991. Το πιο έγινε το Φεβρουάριο φέτος όταν 7 μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφτηκαν το Σίδνεϊ, την Καμπέρα και την Αδελαίδα. Αυτό που μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα ως αντιπροσωπείας ήταν να ακούσουμε παντού το πώς η Αυστραλία μετατοπίζει την εστίαση της σε μια δυναμική εξωτερική πολιτική προς την Ασιατική Ήπειρο λόγω του εξαιρετικά μεγάλου δυναμικού της Ήπειρου αυτής. Ε, ενώ η άποψη για την Ευρώπη αυτή που ακούσαμε τουλάχιστον έλεγε ότι είμαστε οπισθοδρομικοί αρτηροσκληρωτικοί και ότι χάνεται το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ήπερο. Έτσι λοιπόν ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ψάχνετε νέες αγορές, αναζητείτε νέα δυναμική σχέση με, την, ε, με τις χώρες της ε, Ασίας. Αυτή η σχέση Αυστραλίας-Ασίας δεν θα πρέπει πιστεύω να διακυβεύσει ή να υπονομεύσει την παραδοσιακή στενή σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ε, δεν υπάρχουν μόνο αυτές ε, οι περιοχές του κόσμου, αλλά υπάρχει και ο ειρηνικός. Ας μην ξεχνάμε ότι 650 650.000 Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς δεν είναι ορατή η παρουσία της, ε, των Ευρωπαίων πολιτών και η δύναμή τους σε αυτή την περιοχή. Μήπως θα μπορούσε η Αυστραλία να βοηθήσει σε στενότερη συνεργασία και γεωπολιτική συνεργασία με τις χώρες του Ειρηνικού, τα νησιά του Σολομόντα, Φίτζι και Ανατολικό Τιμόρ. Η Αυστραλία το 2013 και το 2014 θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ε, στην ηγεσία της ομάδας G20 και θα ήθελα να ξέρω ως υπουργό Εξωτερικών ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι σε αυτή τη διετή συνεργασία. Ο κύριος Μπροκ, ο πρόεδρος έχει τόσα ερωτήματα να απαντήσει ο Πρόεδρος, να απαντήσει καταρχάς και μετά θα δώσω το λόγο σε άλλους τέσσερις συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας θα εστιάσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στην εδραίωση της ε, ειρήνης στα νησιά του Σολομόντα, ε, στο Ανατολικό Τιμόρ μετά την καταστροφική, τον καταστροφικό εμφύλιο, την διαμάχη. Επίσης, ε, στοχεύουμε και στην ενίσχυση της ειρηνευτικής προσπάθειας στην Αφρική ε, μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας βεβαίως του ΟΗΕ, το οποίο ε, απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ειρήνευσης στην Αφρική. Ε, όσον αφορά τώρα ε, τη συμμετοχή μας στο, στην ομάδα G20 θα ασχοληθούμε με την εργασία, αγορά εργασίας και απασχόληση ιδιαίτερα. Το συζήτησα αυτό εχθές και στη συνεργασία μας θα κάνουμε μία ανάλυση της κατάστασης. Θα ενισχύσουμε τις, ε, τις άμεσες ενισχύσεις βεβαίως της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στην περιοχή της Αφρικής ε, και του Ειρηνικού και θα συμμετάσχουμε και εμείς. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Τάνοκ, θα ασχοληθούμε καταρχάς με τη Συμφωνία πλαίσιο ε, που πιστεύουμε είναι η καλύτερη μέθοδος να προχωρήσουμε με την ε, Ταϊουάν. Για την Ινδία ε, κάνουμε μια διαβούλευση για τις εξαγωγές ουρανίου και θέλουμε να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα της εξαγωγής ουρανίου από τα ορυχεία της Αυστραλίας προς την Ινδία. Είναι στρατηγικά θέματα αυτά από το Φίτζι μέσω του Ινδικού ωκεανού προς το Ιράν υπάρχει μία ροή, μία ροή και θέλουμε να, οι διαβουλεύσεις μας αυτές να είναι τριμερείς. Η Ινδονησία, Ινδία, Αυστραλία, παραδείγματο χάρη σε βέστητα. Και υπάρχει μία συμφωνία πλαίσιο με το τιμόρ μια συνθήκη συνεργασίας η, η οποία έχει ωφελήσει πάρα πολύ το ανατολικό τιμόρ. Συμφωνία συνεργασίας και ενίσχυσης με το Ανατολικό Τιμόρ. Έχουμε επίσης και μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με την Οδυσσία στο θέμα της ε, αντιτρομοκρατική βάση. Έχουν ε, καταδικάσει επί τη βάση της συνεργασίας μας 400 τρομοκράτες. Έχουμε αστυνομικές δυνάμεις που συνεργάζονται με την ε, αστυνομία της Ινδονησίας και μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ινδονησίας είναι ότι κατάφεραν να δραστηριοποιηθούν εντονότατα σε αντιτρομοκρατικές ε, ε, ε, εκστρατείες, σε αντιτρομοκρατικά προγράμματα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στον Παλί. Τώρα, Κίνα και Βόρειος Κορέα. Αναγνωρίζουμε το πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο έχει παίξει Κίνα στο να αναχαιτήσει, αναχαιτήσει την πολεμοχαρή στρατηγική της Βορείου Κορέας. Ε, πιστεύω ότι η Κίνα δεν μπορεί να μας αποκαλύψει όλες τις σχέσεις και τις πτυχές ε, ε, διαβούλευσης με τη Βόρειο Κορέα, αλλά χαίρομαι διότι έχει αναλάβει ένα θετικό ρόλο η Κίνα. Αυτό το θέμα στην Νότια Ανατολική σημασία των φορολογικών παραδείσων έχει πραγματικά αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και Ένα μέτρο το οποίο θα προωθήσει τη συνεργασία με την Κίνα θα είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου. Πιστεύω ότι η νέα ηγεσία το έχει αναγνωρίσει. Εάν θέλουμε πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία και ο Βίντζαου Τζαουμπάου και ο Πρωθυπουργό Λί έχει πει, έχουν δηλώσει ότι πρόοδο σε αυτά τα δύο ζητήματα θα επιτευχθεί μέσω τη εδραίωση του κράτου δικαίου. Κάθε φορά που αναφέρουμε τι ανησυχίε και τι επιφυλάξει μα, ο Πρωθυπουργό Λί μα λέει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Ε, μου το λέει έτσι με με μία προσέγγιση, με έναν τρόπο που με κάνει να πιστεύω ότι θα υπάρξει και περαιτέρω πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και δέσμευση της νέας ηγεσία στη μετάβαση στο κράτος δικαίου και στις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις όπως τη ζήτησε η Παγκόσμια Τράπεζα. Όσον αφορά τώρα τον ε, χειρισμό της μειονότητας των Ροχίνγκα στην, ε, στο Μιανμάρ, Μίλησα με εκπροσώπους, επισκέφθηκα την κοινότητα των Ροχίνγκας στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα και πιστεύω ότι είναι ε, μία μεγάλη πρόκληση η κατάστασή του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η, η ο χειρισμός τους στο Μιανμάρ έχει ιστορία δεκαετιών. Δηλαδή οι προκαταλήψεις τους είναι ριζωμένες βασιά στη συνείδηση ε, του Μιανμάρ. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις συζητήσεις, να πιέσουμε έσως μέχρι ότου διαπιστώσουμε ότι γίνεται πρόοδος και στο χειρισμό των άλλων μειονοτήτων και των Ροχίνγκας, ειδικά που υποφέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό ακριβώς θα πιέσουμε, θα συζητήσουμε και θα επισκεφθώ τον Ιούνιο τα στρατόπεδα προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί. Το, την Παρασκευή στο Σίδνεϊ θα έρθει ο Υπουργό Εξωτερικών του Ανατολικού Τιμόρ και δεδομένου ότι είναι μια πολύ μικρή και φτωχή χώρα ε, θα παίξει ουσιαστικό ρόλο η συμφιλίωση με την Ινδονησία. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να εκπονήσουμε ε, σχέδια συνεργασίας και συμφιλίωσης μεταξύ Ανατολικού Τιμόρ και Ινδονησίας. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν δεσμευθεί. Δεδομένου ότι υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος ε, στόχος να ε, συμπράξει, να συμμετάσχει στο ΑΣΕΑΝ το Ανατολικό Τιμόρ. Όταν, όταν εντάχθηκε το Λάος στο ΑΖΕΑΝ, θέλουμε να ακολουθήσουμε και εμείς την ίδια οδό, διότι αυτό ήταν επιτυχές τότε. Πιστε... Όσον αφορά την Ταϊουάν, πιστεύουμε στην ενία, σε μία Κίνα και αναγνωρίζουμε το θετικό ρόλο της, των ΗΠΑ και της διπλωματίας. Αναγνωρίζουμε την συνετή στάση, ας πούμε, την, ε, που, που, που έχει δείξει η ηγεσία του, της Ταϊουάν. Η Ταϊουάν ήταν ε, επαρχία της Κίνας ε, μέχρι ότου κατελήψει από τους Ιάπωνες στον Κινέζικο-Ιαπωνικό πόλεμο. Εμείς ποτέ δεν έχουμε αλλάξει την άποψή μας ότι είναι ήταν επαρχία και της Κίνας και ζητούμε την ε, ειρηνική επανασύνδεση της Ταϊουάν με την Κίνα. Έχουμε παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατείας. Έχουμε ε, μία βάση στον αραβικό κόλπο. Ο Ζαν Κλόντ Αντάμ, πρωθυπουργός των Σεχελών, μου είπε ότι η χώρα του έχει χάσει ένα τρίτο της, ε, της ετήσιας προμήθειας καυσίμων λόγω της πειρατείας, διότι έχουν απαγάγει τα πετρελαιοφόρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος της καταστροφής ζημιάς. Έχουμε λοιπόν δεσμευθεί πολύ έντονα και έχουμε συνεργαστεί μαζί σας σε όλο το, την περιοχή του, στο κέρα της Αφρικής για ε, την καταπολέμηση της πειρατείας. Τώρα για την κινέζικη εξωτερική πολιτική, οι Κινέζοι πρέπει να αξιολογήσουν την κατά πόσον θα είναι συνεργάσιμη ή όχι μετά το 2008 στις διενέξεις που υπάρχουν για τη, στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι διατάξεις του δικαίου της ε, θαλάσσης και του διεθνούς δικαίου. Και ενθαρρύνουμε την εργασία που έχει κάνει το ΑΣΕΑΝ προς έναν ε, κώδικα ε, δεοντολογίας. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχουν ιστορικά, ένα ιστορικό παρελθόν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, σχεδόν δηλαδή, η αιτία του ήταν το περιστατικό στην Ταγκέρη ε, χρόνια πριν από το 1914 και επίσης μία ε, μία ιστορία της Ευρώπης δείχνει ότι υπήρχε ε, διένεξη και σύγκρουση στη θάλασσα πριν αρχίσει ο πόλεμος στη στεριά. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε την Κίνα να ακολουθήσει αυτό τον κώδικα διοντολογίας αυτές τις ε, διενέξεις της, νότιας θάλασσας. Η, η μία είναι δεοντολογία για την ε, διεξαγωγή των συζητήσεων και εν συνεχεία δεοντολογία για την ρύθμιση των διενέξεων έτσι ώστε να μπορούν να συνυπογράψουν όλοι και να έχει αξία αυτή η συμφωνία. Η εταιρική μας σχέση με την Κίνα βασίζεται σε αμοιβέ συμφέροντα και ορισμένες αμοιβέ αξίες ε, στην ειρηνευτική ανάπτυξη της περιοχής η δυναμική της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής θα από τη συμπεριφορά τους στη διεθνή σκηνή και από την ενεργό συμμετοχή τους στα, στις, παγκόσμια φόρουμ και στην ενασχόλησή τους με τα παγκόσμια ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για τις πραγματικά εκτεταμένες εκτεταμένες αλλά και ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις που κάνατε για την εξωτερική πολιτική. Επιτρέψτε μου τώρα σε αυτό το δεύτερο γύρο, εδώ βρίσκομαι κύριε Υπουργέ, να σας θέσω δύο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, η οποία, από τις οποίες η μία αναφέρεται πάλι στην Μιανμάρ ως μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλώνω σαφώς ότι συμφωνώ με τις πολιτικές εκτιμήσεις. Το τονίζω αυτό. Όταν θα πάτε στην Μιανμάρ, σας παρακαλώ ωστόσο, να μην ρωτήσετε μόνο τι γίνεται με τους Ροχίνγκας και με την κατάστασή τους ως μουσουλμάνων, να ρωτήσετε και για τους Κατσίν, που είναι χριστιανοί και οι οποίοι βρίσκονται λίγο πολύ στην ίδια θέση στην Μιανμάρ με τους προαναφερθέντες. Παρ' όλα αυτά, σας επενώ για τις πολιτικές σας εκτιμήσεις της καταστάσεως στη χώρα αυτή. Η κυβέρνηση αυτή, στην περίοδο που ασκεί την εξουσία, κατάφερε πολλά. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την αντιπολίτευση, αλλά στην αντιπολίτευση, έτσι έχω αντιληφθεί πλέον, περιλαμβάνονται πολλές ομάδες οι οποίες κινούνται και νομίζω είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτή την αντιπολίτευση. Χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά. Δεύτερη ερώτηση. Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας εξήγησε τις βασικές γραμμές. Ως μέλος της αντιπροσωπείας αυτής ήμουν τον Φεβρουάριο στην χώρα σας και σας ευχαριστώ εδώ ρητά για την θαυμάσια φιλοξενία αλλά και για τη δυνατότητα που μα δώσατε να συνομιλήσουμε μαζί σας. Έμαθα από εσά ότι η χώρα σας, και αυτό με ενθουσίασε πραγματικά, ρώτησα δηλαδή ποιες γλώσσες, γλώσσες μαθαίνουν τα παιδιά σας. Και η απάντηση που άκουσα ήταν κινέζικα και ιαπωνικά. Πραγματικά έχετε τα μάτια σας στραμμένα στο μέλλον. Πώς διαμορφώνεται ωστόσο τη συνεργασία Αυστραλίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. εννοώ την εμπορική συμφωνία και ιδιαίτερα τον γεωργικό τομέα. Διότι η Ευρώπη είναι ο δεύτερο ή ο τρίτο μεγαλύτερο εταίρο τη Αυστραλία. Η Αυστραλία για την Ευρώπη, ωστόσο, έρχεται σε 15η θέση. Επομένω, μια εμπορική συμφωνία, ιδίω στον αγροτικό τομέα, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την Αυστραλία. Ακούω τώρα ότι ορισμένα θέματα, παρόλο που έχουν προχωρήσει, είναι ακόμη εκκρεμή. Αν κατάλαβα καλά, εσείς θέλετε πρώτα να ολοκληρωθεί η πολιτική συμφωνία και μετά να προχωρήσετε στην εμπορική. Ή μήπως δεν κατανόησα καλά, κύριε Υπουργέ. ο κύριος Πάσκου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για την κατάσταση στην Ευρώπη μετά από τον πρώτο πόλεμο, ή μάλλον πριν από τον πρώτο πόλεμο. Η θεωρία των διεθνών σχέσεων λέει, αν θέλετε ειρήνη στο σύστημα, πρέπει να έχετε ειρήνη στο κέντρο, στο επίκεντρο του συστήματος. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο του συστήματος. Και είχαμε είχαμε για, μεγάλη, για πολλά χρόνια ειρήνη και μετά είχαμε τον πρώτο πόλεμο, διότι οι μονομερείς δράσεις τελικώ υπερίσχυσαν αντί των πολυμερών. Για να φτιάξουμε την ειρήνη, δώσαμε στους εαυτούς μας δύο πολυεθνικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί κατήσχησαν στις πολυμερείς σχέσεις μας. Αν έχει κανείς τη δυνατότητα τώρα να μπει στο κέντρο του συστήματος, και να ενισχύσει και να ενθαρρύνει τον, την πολυμερή σχέση έναντι των μονομερών δράσεων. Ευχαριστώ σε Ρόμπερτ Άτκινς. Χαίρομαι που σας βλέπω, κύριε Υπουργέ. Ωραία που βλέπουμε και κάποιον από τους αντίποδες που έρχεται και μας μιλεί. Τέσσερα ερωτήματα. Πρώτο, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της κινέζικης δηλώσεως ότι θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις ώστε να είναι πιο δραστήριε ό,τι αφορά την προστασία των κοινωνικών συμφερόντων, κατά πάσα πιθανότητα στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά όχι μόνο. Δεύτερο, ποιε θα είναι οι επιπτώσει επί τη δραστηριότητα τη Αυστραλία για την διατήρηση τη ειρήνη, είτε ό,τι αφορά τον προπολογισμό σα, είτε στο τι θα επαγρυπνείτε, για ποιο πράγμα θα επαγρυπνείτε κλπ. Ε, ε, τρίτο, άλλο θέμα. Ποιε θα είναι οι επιπτώσει, άλλο θέμα τώρα. Ορισμένα από τα νησιά του Νότιου Ειρηνικού υφίστανται μεγάλη βλάβη λόγω της αύξησης της στάθμης των υδάτων και η Αυστραλία διαθέτει κονδύλια από το προπολογισμό τη για να βοηθήσει τα νησιά αυτή. Μπορείτε να μα πείτε λίγο περισσότερα πράγματα. Το πιο σημαντικό στο ερώτημα που έχω για σας και που δεν έχει βέβαια καμιά εύκολη ε, απάντηση πριν από το τέλος του καλοκαιριού είναι ποιο θα κερδίσει στα λεγόμενα ashes, δηλαδή στο κρίκετ μεταξύ Αυστραλών και ε, των υπολείπων χώρων τη κοινοπολιτεία. Πόσελτ, χωρί μικρόφωνο. Τώρα με μικρόφωνο. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσει, κύριε Υπουργέ. Πρώτη, Ινδονησία, Φιλιππίνες. Για τις Φιλιππίνες δεν μιλήσατε. Μεγάλα νησιωτικά κράτη με σημαντικές αποσχιστικές κινήσεις. Η εικόνα που περιγράψατε ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη για την Ινδονησία. Πώς κρίνετε αυτές τις αποσχιστικές κινήσεις στις δύο μεγάλες αυτές νησιωτικές χώρες. Βλέπετε να είναι αυξανόμενος κίνδυνος ή μειούμενος. Δεύτερη ερώτηση. Σχετικά με χώρα με την οποία συνδέεται ιδιαίτερη η Αυστραλία. Παππούα Νέα Γουινέα. Πώς κρίνεται εκεί τη σταθερότητα και το μέλλον της Παππούα Νέα Γουινέα. Θαυμάσεις πάλι οι ερωτήσεις που μου θέσατε. Βέβαια δεν επιτρέπεται να ξεχνούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη Μιανμάρ. Συμφωνώ με την ε, παρατήρηση σας για, το, για τους Κατσίν. Περιλαμβάνουμε ε, τα θέματα αυτά στη συζήτηση γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση για την Μιανμάρ είναι όχι μόνο η οικονομική ε, ανάπτυξη για μια πολύ φτωχή χώρα αλλά και η συμφιλίωση. Εμείς συμβάλλουμε εκεί σε διάφορα προγράμματα συμφιλίωσης. είμαστε και οι μεγαλύτεροι δωρητές. Ε, συνεργαζόμαστε εκεί με το Ενωμένο Βασίλειο. Έχουμε χτίσει ένα σχολείο έξω από τη Ρανγκούν. Εκπαιδεύσαμε και τους δασκάλους, προσφέραμε και τον εξοπλισμό. Βγαίνοντας από το σχολείο, με πολλούς υπερήφανους γονείς γύρω που έβλεπαν τα παιδιά τους, βέβαια μια μέρα όπου που ε, είχε πάει ο Αυστραλός Υπουργός των Εξωτερικών και ένας από τους γονιούς φορούσε ένα ε, t-shirt που έλεγε υπέρ της δημοκρατίας. Και είπα εγώ, είδα την Αούν κι χθε. Α, ναι, και εγώ την είδα τηλεόραση. Ε, αυτά τα δείχνουν τώρα και στην τηλεόραση την επίσκεψη του Αυστραλού Υπουργού Εξωτερικών σε αυτή την ε, εικόνα της αντιπολίτευσης που είναι η Αμοσονική. Είναι μια χώρα η οποία τώρα έχει ρηχτεί να φτιάχνει σχολεία, να στηρίζει τους νέους της και η Ευρώπη και η Αυστραλία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συμβάλει ώστε να γίνει ιστορία επιτυχίας και η Μιανμάρ να μπει σε μια ζώνη ευημερίας μεταξύ Ασάμ και Ιουνάν. Και υπάρχει προοπτική οικονομικής ανάπτυξης που θα προσφέρει δυνατότητες στους ανθρώπους αυτούς και που μειώνει και την σημασία αυτών των διαφορών όπως με τους Ροχίνικα και τους Κατσίν. Η συνεργασία για, με την Ευρώπη για την ανάπτυξη της Ασίας θεωρώ ότι υπάρχουν αξίες που έρχονται από την Ευρώπη. Οι αξίες μας είναι ευρωπαϊκές. Ο λόγος για τους οποίους έρχονται οι ήρθαν οι μετανάστες στην ε, Αυστραλία είναι το πολυφωνικό μας σύστημα. Καθιστά την Αυστραλία ελκυστική για μετανάστες από την Ινδία ή την ε, Κίνα. Πέρασαν πολλά δεινά για να φτάσουν στην Αυστραλία διότι αναζήτησαν την ελευθερία που προέρχεται από τις ευρωπαϊκές αξίες και που αυτές, σε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες χτίστηκαν και οι Αυστραλιανοί θεσμοί. Ο Σερόμπερτ Ρόμπερτ με, ρώτησε για, για τον εξυγχρονισμό. Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας θα ακολουθηθεί και από τον εξυγχρονισμό των κινέζικων στρατιωτικών δυνάμεων. Οι Κινέζοι πρέπει να φροντίσουν να μειώσουν τους φόβους που τους προκαλεί αυτό με το να είναι διαφανής. Είπαμε στους Κινέζους, προωθείτε τον εξυγχρονισμό των δυνάμεών σας, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και τη συνεργασία μας με τους συμμάχους μας και ιδίως τις Ενωμένες Πολιτείες. Για τον ειρηνικό μου βάλατε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Όσοι γνωρίζουν, όσοι θέλουν να μάθουν περί κλιματικής αλλαγής πρέπει να πάτε στο Κιουραμπές μαζί με τον πρόεδρο που δεν είναι νησιωτική χώρα, είναι ατόλη. Ένα κράτος πάνω σε μια ατόλη. Είχαμε ένα δρόμο που θέλαμε να φτιάξουμε. Από τη μια μεριά είναι ο ωκεανός και σηκώνεται η στάθμη του νερού. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό μολύνει τα υπόγεια ύδατα. Το πόσιμο νερό δηλαδή. Κάνουμε λοιπόν δημόσια έργα για να αναστείλουμε την ημερομηνία όπου θα αναγκαστεί ο πληθυσμός της ατόλης Κυριμπάτη που είναι 100.000 να σηκωθούν να φύγουν, να εγκαταλείψουν το νησί τους. Τους εκπαιδεύουμε σε, ως μηχανικούς στα ηλεκτρονικά κτλ. με επίπεδο αυστραλιανό, ώστε όταν θα φύγουν από την ατόλη τους να μπορούσαν να έλθουν όχι ως πρόσφυγες, αλλά ως υπερήφανοι μετανάστες. Πήγα σε ένα τεχνικό κολέγιο που χρηματοδοτούμε, όπου οι νεαροί αυτοί μαθαίνουν αγγλικά και μαθαίνουν και τη δουλειά σε αυστραλιανό επίπεδο. Όμως η κλιματική αλλαγή θα αναγκάσει ανθρώπους με χιλιετή ε, πείρα στο πώς να χειρίζονται τα πλούτη του ωκεανού να εγκαταλείψουν τα νησιά τους. Αυτοί έχουν μεικτό αίμα από Μαλαισιανούς και Ευρωπαίους. Όλα αυτά πρέπει να τα εγκαταλείψουν και θα εξαφανιστεί ο πολιτισμός αυτός λόγω της θέρμανσης του πλανήτη. Τα βλέπετε αυτά τα πράγματα στο Κυριμπάτι και βλέπετε ότι το νερό ανεβαίνει. Εσείς κύριε Πόσελτ, θέσατε ενδιαφέροντα ε- ερωτήματα για τα αποσχιστικά κινήματα στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες. Η Μαλαισία βοήθησε, συνέβαλε, διαμεσολάβησε στην σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ισλαμιστών ε, αυτονομιστών στις Φιλιππίνες και της κυβέρνησης που υπόσχεται πολλά. Στην ίδια την Ινδονησία πιστεύουμε ότι ένα μέτρο της επιτυχίας τους θα είναι ο τρόπος που θα χειριστούν τα αποσυστικά κινήματα στο Άτσε. Εγώ μίλησα με τον, με ε, ε, πρωθυπουργό του πριν από ένα μήνα και ο ίδιος έθεσε το θέμα της Παπούα και μίλησε για την δέσμευσή του για την χορήγηση ειδική αυτονομίας στην επαρχία αυτή. Η Αυστραλία δέχεται την ε, Ινδονησιακή κυριαρχία επί των επαρχιών της Παπούα και ενθαρρύνουμε τους φίλους μας να προχωρήσουν στη δημιουργία του ειδικού καθεστώτος αυτονομίας που αναπτύσσονται και θα μειωθεί η διαφορά στο επίπεδο ευημερίας. Παππού Ανέγου, είναι εκεί ενθαρρυνόμαστε ιδιαίτερα από την ε, ηγετική ικανότητα του Πρωθυπουργού σε κοινοβούλιο 111 μελών έλαβε πλειοψηφία 90 ε, ψήφων. Προχωρεί σε ένα πρόγραμμα ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και ε, βελτίωση της υγείας των πολιτών του. Πολύ φτωχή χώρα, με μεγάλη εθνοτική ποικιλία, με πολύ δύσκολη τοπογραφία, ωστόσο έκαναν πέρσι δημοκρατικές εκλογές και επέτρεψαν του κόσμου να πάει στις κάλπες και να εκλέξει τους ε, αντιπροσώπους του. Εφόσον η Παππούα Νέα Γουινία μπορεί να κάνει ελεύθερες εκλογές, με ελευθερία του συνεταιρίζεστε κλπ. Τότε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μπορεί να διεξαγάγει ελεύθερες εκλογές. Σημαντικό επίτευγμα, υπερήφανο επίτευγμα λοιπόν του, της Παππούα Νέα Γουίνια. Τώρα για τις Ashes. Εγώ δεν είμαι τόσο φανατικός οπαδός. Εδώ ο πρέσβης μου μου λέει όμως η ιστορία έχει δείξει την διαρκούσα υπεροχή των ομάδων κρίκετ των Αυστραλών απέναντι στις Βρετανικές. Και πιστεύουμε ότι αυτή η υπεροχή θα διατηρηθεί. Πολύ διπλωματική απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή και που κάνατε και την συζήτηση και τις παρατηρήσεις σας. Να θυμίσουμε στην Αυστραλία ίσως ότι και η Ευρώπη παίζει ακόμα ρόλο, όπως παίζει και η Αυστραλία και όχι μόνο λόγω των πρώτων υλών. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε συμφωνία πλαίσιο να ολοκληρωθεί το σύντομο το δυνατό μόλις πήρε ένα μήνυμα ότι ο Γενικός Κυβερνήτης σας θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες με μια επιχειρη... αντιπροσωπή επιχειρηματιών για να συζητήσουμε περισσότερο τα θέματα αυτά στην 1η Ιουλίου. Κάτι που δείχνει ότι η διαδικασία είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία μας ε, θέτουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο τη συνεργασία με την Αυστραλία. Και ότι εδώ εξετάζουμε τη συνεργασία μας με την Ασία και από την οπτική γωνία των συμφερόντων αλλά και από εκείνη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πιστεύω ότι οι κοινέ αξίε που και οι δύο πλευρέ έχουμε θα πρέπει να μα οδηγήσουν να έχουμε ακόμα στενότερη συνεργασία με τη μεγάλη χώρα της Αυστραλίας και μεταξύ μας. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.